Ora, l'ordine del giorno. Στην ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού και ξεκινούμε με τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ελλάδα καταβάλει το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη ε, μνημειώδη προσπάθεια παράλληλα με την οικονομική σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει σε ένα περιβάλλον ακραίων και ρατσιστικών φωνών. παρ' όλα αυτά χειροπιαστά αποτελέσματα ήδη βλέπουμε με τις προσπάθειες που γίνονται. οι ροές των παρανόμων μεταναστών στον εύρο έχουν μειωθεί κατά πολύ και συνολικά οι ροές στη χώρα μας έχουν περιοριστεί λόγω της καλύτερης φύλαξης των συνόρων ε, και θυμίζω ότι την περίοδο αυτή η χώρα δέχεται μεγάλη πίεση και από τη συρία. είναι όμως η περίοδος και γι' αυτό το αναφέρω αυτό να αντιληφθούμε ότι πλέον τα βάρη της παράνομης μετανάστευσης δεν μπορεί η ευρώπη να τα σηκώσει από μόνη τη. είναι η ώρα τώρα να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τη ρήτρα κατανομής που ήδη έχουμε συμπεριλάβει σε μη νομοθετικά κείμενά μα. η ιδέα αυτή μπορεί να είναι το καλύτερο δυνατό εργαλείο για τη συνέχεια ένα εργαλείο που θα επιτρέψει στην ευρώπη να λειτουργήσει με την πραγματική αλληλεγγύη και την ισότιμη κατανομή των βαρών που χρειάζεται. σας ευχαριστώ πολύ. Το 2009 ισχυρό σεισμός έπληξε την περιοχή Εμπρούζο στην Βόρεια Ιταλία. Δεκάδες ανθρώπινα θύματα, καταρρεύσεις κτηρίων, σχολείων, νηπιαγωγείων, νοσοκομείων και πολλών ε, υποδομών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακάπτοντας ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες και μετά από πρόταση Ιταλών συναδέλφων μας, ε, κινητοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και ενέκρινε το ευρωκοινοβούλιο 500 εκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση των κατοίκων των σεισμοπαθών και την ε, αποκατάσταση των ζημιών. τρία χρόνια αργότερα μόλις την περασμένη δευτέρα κυρία πρόεδρε ιταλικό δικαστήριο ε, καταδίκασε έξι συναδέλφους σεισμολόγους επειδή δεν πρόβλεψαν το σεισμό. η απόφαση αυτή είναι παράλογη η απόφαση αυτή είναι πρωτάκουστη και κατά τη γνώμη μου επικίνδυνη η απόφαση αυτή δεν καταδικάζει τους σεισμολόγους δεν καταδικάζει τους επιστήμονες καταδικάζει την ίδια την επιστήμη και όλες τις επιστήμες. δεν είναι πρόθεσή μου να ζητήσω από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο παρέμβαση στην ανεξάρτητη ιταλική δικαιοσύνη αλλά επιτρέψτε μου κυρία πρόεδρε να πω ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. ευχαριστώ πολύ. President, Η κυρία Τέιλορ. Ε, κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί ε, ε, βουλευτές, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέτηση του κυρίου Ντάλι. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που πολλοί από εσά διάβασαν στα ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση. Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι πολλά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί ακόμα και το εάν είναι τελικά ένοχο ο κύριο ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τέτοια θέματα και ελπίζω αυτό να γίνει στο μέλλον. Πιο σημαντική η οχι δεν ειναι σαφες οι οι ευρωπαιοι πολιτες θα πρεπει να ενημερωνονται καλυτερα σχετικα με τετοια θεματα και ελπιζω αυτο να γινει στο μελλον πιο σημαντικη η ανησυχία είναι ε, το, η κατάσταση με την ε, οδηγία ε, για τα προϊόντα καπνού μετά την παρέτηση του κυρίου Ντάλη. Είναι το, το ο καπνός σκοτώνει πολλούς κάθε χρόνο και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η Κομισιόν λέει ότι δεν θα καθυστερήσει η οδηγία και ότι θα συνεχίσουν μόλι ε, υπάρχει νέος Μαλτέζο επίτροπο, αλλά αυτό μπορεί να κρατήσει μήνε. Ε, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχει ολοκληρώσει τι εργασίε πάνω, ε, πάνω στην οδηγία και από ό,τι κατάλαβα έχει ολοκληρωθεί η διοργανική συνεννόηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να υπάρχει νέος Επίτροπος προτού να προωθηθεί αυτή η νέα οδηγία. Καλώ την Κομισιόν να δημοσιεύσει γρήγορα την πρόταση αυτή προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, σας ε, πω κάτι που βρήκα στο YouTube ε, πριν κάποιου μήνε. Κάποιο έλεγε ότι «Μ' αρέσει το τραγούδι αλλά δεν μ' αρέσουν τα ε, πειρατικά βίντεο». Συγγνώμη λοιπόν ε, όσον αφορά το copyright. Αυτό δείχνει ακριβώ ποιο είναι το πρόβλημα το copyright. Ε, όταν ένας ε, χρησιμοποιεί τα πολιτιστικά αγαθά με τον τρόπο που βρίσκει πιο φυσικό. Υπάρχει λοιπόν ε, ένας DJ που λέγεται Gucci και έχει φτιάξει ένα μουσικό βίντεο ε, το οποίο ε, είχε εμπνευστεί από την σειρά Game of Thrones που βασίζεται σε μια σειρά βιβλίων του George R. R. Martin. Εμένα μου προκάλεσε έκπληξη το βίντεο αυτό επειδή ο χρήστης σχολιάζει τη δική του συμπεριφορά και δείχνει ακριβώ την αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που θέλει να κάνει και τους κανόνε για το ε, copyright και δείχνει ε, πώς ε, τελικά οι κανόνε του copyright επηρεάζουν την καθημερινή ζωή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάφτον. Uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κάποιο ε, το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο πρώην Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να αποκεντρωθεί, ενώ ο Πρωθυπουργό είπε ότι εάν ε, ε, επιτύχουν τα μέτρα για την Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να γίνουμε ομοσπονδία. Ο Ντέιβιτ Κάμερον είπε ότι θα γίνει δημοψήφισμα για οποιαδήποτε νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη μετά την ε, ε, προηγούμενη Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Τώρα λοιπόν ο κύριος Μπαρόσο ζητά να έχουμε μία συνθήκη που θα έχει δημοκρατικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς θέλουμε να ξέρουμε αν θα έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει. Πότε θα γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Το UKIP ε, θα βγει στην κορυφή στις επόμενες εκλογές. Γιατί να μην δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να επιλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το 2013. Αν η Ευρώπη θέλει να γίνει ομοσπονδία ε, και θέλει να συγχύσει τα πράγματα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει τη συζήτηση για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μεστσάρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2004 δέκα νέε χώρες ε, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ακολούθησε συζητήσεις για ε, θέματα προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένου και του θέματος των διαταγμάτων Μπένες ε, που επέτρεψε να παραμείνουν οι διακρίσεις νόμιμες ε, σε αυτήν ε, την χώρα που είναι όνειδος εθνοκάθαρσης. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα διατάγματα αυτά δεν έχουν νομικές επιπτώσεις σήμερα διότι τα δικαστήρια τα χρησιμοποίησαν για ορισμένες υποθέσεις. Κατά την προσχώρηση ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δεκτό ότι δεν επρόκειτο τα διατάγματα αυτά να είναι εμπόδιο, αλλά είναι εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνηγορεί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ερευνήσει για τις νομικές αντιφάσεις που απειλούν τις μειονότητες της Ευρώπης που πρέπει να τύχουν ίσης μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουσέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία διότι κάποια κράτη-μέλη... Α, συγγνώμη. Δεν είναι η σειρά μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις πολιτικές εξελίξεις στη Μάλτα τους τελευταίους μήνες. Το 2008 το Εθνικιστικό Κόμμα κέρδισε τις εκλογές με 53% και τους τελευταίους αυτούς μήνες έχασε την πλειοψηφία της γιατί είχε μόνο ένα μέλος ε, διαφορά ε, και αρκετά μέλη και του ίδιου του κόμματος καταψήφισαν την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα που ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση δεν έχει σταθερή πλειοψηφία στη Βουλή και χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία, δεν υπάρχει σταθερότητα και μέσα στο κόμμα της. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χειραγωγούνται από το ε, κόμμα που διαθέτει την κυβέρνηση και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε νέες εκλογές ε, και να ακουστεί η φωνή του λαού. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον κρίσης. Χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση και μια σαφή φωνή. Κάνουμε έκκληση λοιπόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει τι συμβαίνει στη Μάλτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ότι ήθελα να καταγγείλω το γεγονό ότι κάποιε κυβερνήσει κρατών μελών ζητούν από τι αστυνομικέ δυνάμει ε, στι διαδηλώσει κατά των περικοπών που γίνονται κυρίω στι νότιε χώρε τη Ευρώπη να δράσουν με βίαιο τρόπο. Καταγγέλλεται λοιπόν αυτή η κατάσταση στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Στην Ισπανία διαθέτουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα οι πολιτικοί θύνοντες ε, και οι δυνάμεις της τάξεως ε, δρούν χωρίς ε, να υπάρχει αναγνώριση όπως προστάζει ο νόμος. Επειδή λοιπόν δεν ε, δηλώνουν ποιοι είναι, οποιαδήποτε ε, παραβίαση, οποιαδήποτε ε, πράξη βίας κατά των πολιτών μένει ατιμωρήτη διότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος είναι. Υπάρχει πολιτική ευθύνη λοιπόν, δεν είναι ευθύνη της αστυνομίας αλλά είναι ευθύνη αυτών που δίνουν διαταγές να γίνονται τέτοιες πράξεις. Επομένως δεν θα πρέπει να μείνει καμία πράξη ατιμόρυτη από τις δυνάμεις της τάξης. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Η χώρα των Βάσκων έχει ένα ε, μοντέλο ανάπτυξης που μαζί με τις ε, πολιτιστικές και κοινωνικές της ιδιαιτερότητες τις κάνει σήμα κατά το θέν. η χώρα των Βάσκων. Εδώ και 30 χρόνια ήμασταν ερήπιο σε βιομηχανικό επίπεδο. Σε 30 χρόνια καταφέραμε να δεκαπλάσιάσουμε το ΑΕΠ μας και φτάσαμε στο επίπεδο της Ολλανδίας. Οι εργασίες και δεσμεύσεις της κοινωνίας των Βάσκων και οι πολιτικές της που υποστήριξαν την πραγματική οικονομία όπως έκανε το Παρτίδο Νασιολίστα Βάσκο που κέρδισε και τις εκλογές την περασμένη Κυριακή κατάφερε να εδραιώσει τη θέση μας και θα καταφέρουμε να πατάξουμε και την τρομοκρατική δράση της ΕΤΑ. Σήμερα ε, μπορούμε να ε, προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να στηρίξουμε τη βιομηχανία, την απασχόληση, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και θέλουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη με ανθρώπινη ανάπτυξη. Θέλουμε να φέρουμε αυτό το ε, θέμα στην Ευρώπη και να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Οι άνδρε και οι γυναίκε ε, τη χώρα των Βάσκων είπαν αυτή την Κυριακή ότι θέλουν να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση και την ταυτότητα και να παραμείνουν στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να παραμείνουμε στην Ευρώπη και να ακούσουν οι πολίτε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αγκουράκη. συγκυβέρνηση στην ελλάδα μαζί με τους ξένους συμμάχους της ευρωπαϊκή ένωση και τρόικα κατέληξε στο μνημόνιο 3 μετά από ένα προκλητικό θέατρο δίθεν διαφωνιών σφαγή μισθών και συντάξεων με μειώσει 35% κατεδάφιση κάθε εργασιακού δικαιώματος άγριες περικοπές σε υγεία πρόνοια εκπαίδευση. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν πεταχθεί στον δρόμο χωρίς επίδομα ανεργίας χωρίς καμία κοινωνική προστασία. χιλιάδες είναι οι άνεργοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. στα ναυπηγεία σκαραμαγκά οι εργάτες κάνουν μόλις τέσσερα μεροκάματα το μήνα. τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι το πρόσχημα τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα για φθηνή εργατική δύναμη είναι εδώ και είκοσι χρόνια στρατηγικό στόχο μονοπωλίων και ευρωπαϊκή ένωση και αστικών κυβερνήσεων. η πρόσφατη έκθεση ρομπάι το ομολογεί χωρί περιστροφέ μνημόνια καπιταλιστική βαρβαρότητα σε κάθε κράτο μέλο. φτάνει πια! λαϊκό ξεσηκωμό λοιπόν για να μπει τέρμα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα να οικοδομήσουν οι εργαζόμενοι τη λαϊκή ευημερία με τη δική τους λαϊκή εξουσία πάνω στα ερήπια της εξουσίας των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και της Κομισιόν σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει καταστήσει αδύνατες τις εργασίες σε μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ε, Ρουμανία. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει σταματήσει τη χρηματοδότηση ε, των σχετικών προγραμμάτων ε, και δεν αμφισβητώ την ορθότητα των ερευνών που έχουν γίνει, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η λειτουργία χιλιάδων ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων διακυβεύεται επειδή οι ρουμανικές αρχές εδώ και μήνες ε, δεν ε, πληρώνουν τις ενισχύσεις. Υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις που παίρνουν τραπεζικά δάνεια για τους δύσκολους καιρούς αλλά πολλά χρήσιμα προγράμματα διακυβεύονται. Δεν δεν μας παίρνει λόγω καταχρήσεων των ε, αρχών ε, να σταματήσουν ε, τα προγράμματα για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γιαρόκα. Θα ήθελα να επικροτήσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 9 και 10 ε, Οκτωβρίου τόνισε ότι ε, η ένταξη των Ρώμα είναι θέμα προτεραιότητας και κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης και να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η κρίση ε, στην ε, Ευρώπη έχει επιταχύνει ε, τις ε, τάσεις που υπήρχαν και όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να επιβιώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον Νοέμβριο προσβλέπουμε στην συμφωνία πάνω στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο ελπίζουμε ότι θα φιλήσει τους περιθωριοποιημένους Ευρωπαίους. Η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θα δώσει προσοχή στις ε, κοινωνικά αποκλεισμένες ε, ομάδες ε, και ελπίζουμε ότι θα προωθηθούν οι σχετικές τροπολογίες στο Συμβούλιο ώστε να βοηθηθούν τα 30 εκατομμύρια των Ευρωπαίων που είναι πιο αποκλεισμένοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντανσίλα. Ξέρουμε ότι δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί λόγω της ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ρουμανία η ε, η ε, μισή συγκομιδή δημητριακών έχει καταστραφεί και αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσμενής για την γεωργία. Για να μειωθούν αυτές οι δυσκολίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα, να επιδείξει αλληλεγγύη με τους γεωργούς που βλέπουν ε, την εργασία τους να ακυρώνεται λόγω της ξηρασίας. Οι τοπικές αρχές, οι εθνικές αρχές έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα ταμείο αλληλεγγύης για να βοηθάει τους πληθυσμούς που πλήττονται από πλημμύρες, παραμετός χάρη. Αλλά χρειαζόμαστε και μέτρα για την ξηρασία επίσης, διότι η ξηρασία έχει μεγάλες επιπτώσεις πάνω στους γεωργούς και στη διατροφική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγιάλα. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στην ε, σε πλημμύρες που είχαμε πρόσφατα στην περιοχή μου, στην ε, Αραγών στην Θετάνια, στο Θήκο Βίγες και στην πρωτεύουσα της Αραγών, στη Σαραγώσα. Ε, πλήττονται πέντε δήμοι, ε, πλήχθηκαν ε, δρόμοι, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια με κόστος που εκτιμάται αυτή τη στιγμή ε, κάτι πάνω από τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή που η, κρίση, η οικονομική κρίση και η ξηρασία πλήττουν την περιοχή μου της Αραγών, οι πλημμύρες ε, τους οδήγησαν πλέον σε απελπιστική κατάσταση και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση του ε, Λαϊκού Κόμματος δεν έδρασε ε, με αποφασιστικότητα, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από τα μέο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει οι κάτοικοι της Αραγών να νιώσουν την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Γκάλαγκερ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, έχω υποβάλει ε, έκθεσή μου σχετικά με τον κανονισμό για ε, την ε, μη αηφόρη αλληλεία που επιτρέπεται από κάποια Ο κανονισμός επιτρέπει στην ε, Επίτροπο Δαμανάκη να επιβάλλει σημαντικές κυρώσεις στις χώρες που εφαρμόζουν μη βιώσιμες μεθόδους αλληλείας όπως είναι η Ισλανδία. Η αλληλεία του σκουμπριού. Ε, θεωρείται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2010 προτού ε, ξεκινήσει η υπεραλίευση από την ε, Ισλανδία. Μέχρι τότε είχαμε σχετικά μικρές ποσότητες αλληλείας του σκουμπριού πριν το 2010, όπου η αλληλεία έφτασε 150.000 ε, τόνους ε, που είναι ε, μη βιώσιμα επίπεδα. Όλα αυτά σχετίζονται και με την κατάσταση στην Ιαπωνία. Θα πρέπει λοιπόν η Επίτροπο να αναλάβει άμεση δράση και να εφαρμόσει τι διατάξει που υπάρχουν στον κανονισμό που είχε σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη στο Κοινοβούλιο μα. Ε, και πάλι οι διαπραγματεύσει ε, ε, κατέληξαν σε αδιέξοδο στο Λονδίνο αυτή τη βδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. Ευχαριστώ πολύ. Την περασμένη εβδομάδα στο Βουκουρέστι έγινε μια συζήτηση για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ε, διοργάνωση από το ΕΛΚ και είχαμε εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν εκεί ο Επίτροπος Ταγιάννη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωποι της Ρουμανικής Κυβέρνησης φάνηκε ότι ανησυχούν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ζωτική σημασία. Πολύ συχνά ακούμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, είναι μακριά από τις ανησυχίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επομένως πρέπει και εμείς ως Ευρωβουλευτής αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε ένα πιο εντατικό διάλογο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες τους πάντα ακούμε διαμαρτυρίες ε, για τις συνθήκες ε, που δεν επιτρέπουν ε, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να λαμβάνονται υπόψη ε, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχουν πιο δελαστικές προϋποθέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η, ε, ευρωβουλευτές ε, έχουν ασυλία. Ωστόσο, ε, πολύ ε, συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάρχηση αυτή. Ω ε, εκπρόσωπο τη Βόρεια Ιρλανδία, εργάζομαστε σκληρά πάνω στην επίλυση τη σύγκρουση και ξέρουμε ότι η επίλυση των διαφορών, επίλυση διαμάχη μπορεί να υπάρξει μόνο με την συνομιλία και αν ξεφύγουμε από τι άκαπτε θέσει και την θέση ότι θα πρέπει ο εχθρό μου να δεχτεί τη θέση Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο μα προέκυψε από ε, μια διαμάχη, από έναν πόλεμο και στόχο έχει να προωθήσει την αλληλεγγύη, θα πρέπει χωρίς ε, δισταγμό να ε, αποστασιοποιηθεί από οποιανδήποτε ευρωβουλευτή που ε, να ε, ε, εκφράζει ακραίες θέσεις. Ο Ευρωβουλευτής Γκρίφινς έκανε δηλώσεις καθώς και μηνύματα στο Twitter τα οποία έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων και τίποτα τέτοιο δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την ασυλία των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νικολέσκου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω ζητήσει από την Κομισιόν να υποβάλει στρατηγική για την καταπολέμηση των καταστροφικών ε, συνεπειών της ε, αύξησης των ε, τιμών των σιτηρών η ξηρασία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των σιτηρών, ε, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Ε, ταυτόχρονα, γεωργοί σε όλη ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν ότι μπορεί να μην έχουν αρκετές ζωοτροφές που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών. Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει ότι θα σταματήσει την εξαγωγή ε, σιτηρών ε, από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ε, στο χρηματιστήριο του Σικάγο. Και είναι μια ε, πολύ συγκεκριμένη κατάσταση αυτή. Να μην ξεχνάμε ότι οι τιμέ θα συνεχίσουν να είναι υψηλέ. Το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς θα φτάσουμε σε ιστορικό υψηλό των τιμών και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια γρήγορη στρατηγική για να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό. Όποτε ε, ρωτάμε την Επιτροπή σχετικά με μια τέτοια στρατηγική, λέει ότι χρειαζόμαστε διαφορετικά μέτρα. Ναι, χρειαζόμαστε τέτοια, χρειαζόμαστε όμω και συγκεκριμένε λύσει, σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάνκι. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Ε, ε, απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, Γι' αυτό ε, παρακαλώ να παραμείνουν στην αίθουσα. Το πρωτόκολλο ε, του ε, το πρωτόκολλο του Κιώτο θα λήξει και θέλουμε επιμήκυνσή του μέχρι το 2020. Τα επιμέρους κρατημέλη όπως και η Ουγγαρία έχουν αναλάβει μέτρα. Υπάρχει όμως και η αρχή που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετράει ως ένα κράτος και γι' αυτό η μείωση των εκπομπών αναμένεται από τα κράτη-μέλη, όπως άλλωστε και από την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία έχει δεσμευτεί για το 6%, έχει όμως ε, ε, κάνει μειώσεις στις τάξεις του 25%. Η Κομισιόν δεν επιτρέπει τα αποθέματα αυτά να μεταφερθούν ε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, παρότι Ε, κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο για, τα, για τις χώρες ε, της ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει συγκεκριμένε προτάσεις και θα παρακαλούσαμε να συζητηθούν οι προτάσεις αυτές στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τσικάου. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ανικανότητα της ε, δεξιάς κυβερνήσεως στη Ρουμανία τα τελευταία χρόνια οδήγησε ε, σε ε, δημοσιονομικές προσαρμογές και στην αναστολή τριών προγραμμάτων που χρηματοδοτούσαν τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2010-2011 η Επιτροπή ε, διαπίστωσε ορισμένα ελαττώματα και κενά ε, στα συστήματα ελέγχου ε, και για την ανταγωνιστικότητα. Η αναστολή αυτή ελπίζω να μην μειώσει τα ποσά. Το, η κυβέρνηση έχει δύο μήνες για να διορθώσει ε, την κατάσταση για να διορθώσει, να καλύψει αυτά τα κενά. Ζητούμε πλήρη συνεργασία της Επιτροπής με την σημερινή κυβέρνηση, ούτω ώστε να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση στη Ρουμανία, προγράμματα τα οποία χρειάζονται τόσο πολύ οι Ρουμάνοι. Ο κύριος Όλιουλαντ. Η κυρία Όλιουλαντ. Κυρία Πρόεδρε, ε, σύντομα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, ασχοληθεί με τους ε, τρόπους ε, υπολογισμού για την παραγωγή του σχιστολιθικού αέριου. Ε, και σκοπός είναι να ε, διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα προϊόντα σχιστολιθικού αερίου. Θέλουμε και στο μέλλον να μπορούμε να παράγουμε αέριο καύσιμα από σχιστόλιθο για να μειώσουμε τις εισαγωγές καυσίμων. Το σχετικό σχέδιο όμως θέτει σε δυσμενή καλή θέση στην αγορά ε, τα ε, προϊόντα από σχιστό λιθό. Έτσι όμως ε, δεν πρόκειται να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, του θα αυξηθούν. Και γι' αυτό δεν είναι προς συμφέρον μας η πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή του Νομπέλ είτε έχει κακό χιούμορ ή δεν καταλαβαίνει το θέμα της ειρήνης. Πριν από τρία χρόνια στον Ομπάμα δόθηκε το βραβείο ενώ τρία χρόνια αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας, ε, ένας θεσμός ε, ή μια ομάδα θεσμών δεξιών ε, που ε, έχουν ε, ταξικό πόλεμο σε άλλες τάξεις. Η λιτότητα είναι το όπλο και το όπλο αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο κακοήθη εξ ονόματος των τραπαζιτών, των πλούσιων εναντίον των εργαζομένων ε, σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε, πρέπει λοιπόν να ξαναχτυπήσουμε κι εμείς. Έχουμε τους εργαζόμενους από την Πορτογαλία, την Ισπανία με πολλές διαμαρτυρίες στην Ευρώπη ε, πρέπει να υπάρξει μια γενική απεργία στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Μάλτα και στην Κύπρο στις 14 Νοεμβρίου με διαμαρτυρίες μαζικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης ελπίζω διότι η μέρα αυτή η 14η Νοεμβρίου θα πρέπει να είναι μέρα που οι εργαζόμενοι θα ε, υψώσουν τη φωνή τους κατά της ε, λιτότητας, θα αντισταθούν ε, και θα μπορεί να είναι το ζωτικό επόμενο βήμα άλλων οπεργιών, ούτως ώστε να σταματήσει το πρόγραμμα λιτότητας στην Ευρώπη. Στον κύριο Βίντλερ τώρα έχω δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ε, νομίζω ότι βρίσκεται σε καμπή η Ευρωπαϊκή Ένωση και απειλείται από την κρίση, από τον λαϊκισμό, τον εξτρεμισμό και την ξενοφοβία. Χαιρετίζω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβούλου και τις προσπάθειες της Επιτροπής να διασώσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την Ευρωζώνη. Πρέπει να εστιαστούμε στην υποστήριξη των πολιτών μας διότι στρέφονται οι πολίτες στις κυβερνήσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο πρόβλημα νομιμοποίησεως. Η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενίσχυση του ανήκειν είναι κάτι που πρέπει να προωθηθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Πιστεύω ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξουμε κεντρικό ρόλο σε αυτή όλη τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω λίγο για την ε, διάσκεψη που διοργανώνω εδώ στο Κοινοβούλιο για την ε, παγκόσμια συνεργασία της επιστήμης. Οργανώνουμε ε, μια διοργάνωση στη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας στις 14 Μαρτίου ε, ως τμήμα της Παγκόσμιας Συνεργασίας Επιστήμης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ιρλανδική Προεδρία θα φιλοξενήσουν αυτή την ε, διοργάνωση. Ε, και το σκεπτικό είναι ότι έχουμε μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και όχι ανταγωνισμός και θέλουμε οι επιστήμονες και όσοι χαράσουν πολιτική να συνεργαστούν και ελπίζουμε να έχουμε και εκπροσώπου από 100 χώρε ε, από όλο τον κόσμο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνες τι ε, ημέρε. και αυτό να αποτελέσει τη βάση της συνεργασίας, ώστε να μπορέσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε καταλήλως ε, σε όλες, όλες τις δυνατότητες που αναφέρονται στο Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίρκη απουσιάζει. Ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε επανειλημμένως τον κύριο Νάιτζελ Φάρατς από το UKIP. Έχουμε και την σημαία εκεί πέρα στην ε, κενή του θέση να αναφέρεται στα ε, προβλήματα και την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται όμως με το δικό του το κόμμα. Πριν από δύο χρόνια ο Νάιτζελ Φάρατς ζήτησε απόλυτη διαφάνεια για τις δαπάνες των Ευρωβουλευτών του και ζήτησε κάθε τρεις μήνες να υπάρχει μια δήλωση των δαπανών τους. Αλλά και πάλι το UKIP ε, ψευδόταν ασύστολα. Δείτε την ιστοσελίδα τους. Οι δαπάνες ε, αποτελούν αποχήμα της φαντασίας που αναφέρονται εκεί στο στο σελίδα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και όλα είναι πλασματικά στοιχεία. Ε, το UKIP τώρα έχασε τα, τα έσοδά του και επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των οικονομικών του και αυτοί έχουν χάσει τις αποδείξεις τους. Ο αναπληρωτής του, ο Πολ Νάτολ, δεν έχει επικαιροποιήσει τους λογαριασμού του εδώ και δύο χρόνια. Οι πληροφορίες είναι κάποιες γενικές δαπάνες, αλλά αναφέρονται σε ένα κλάσμα μόνο των όσων γνωρίζουμε ότι πληρώνονται οι ευρωβουλευτές. Πού είναι τα υπόλοιπα πηγαίνουν, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των ευρωβουλευτών. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάλλιστα να υποθέσουμε ότι πήγαν στην τσέπη του, εκτός και αν μπορεί με κάποιο τρόπο να μας εξηγήσει τι απέγιναν αυτά τα χρήματα. Το UPKIP λοιπόν δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Πρόκειται για ένα βρώμικο κόμμα το οποίο ε, παριστάνει ότι είναι αθώο και έντιμο και την επόμενη φορά που θα έρθει εδώ ο κύριος Φάρατς και θα θέσει ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα περισσότερα μέλη θα πρέπει να ζητήσουν απαντήσεις από αυτόν. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, περατώθηκε η συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο, ο οποίος ε, έμεινε εδώ μέχρι το τέλος της συζήτησης.